Για την λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν δεν διαφωνούμε με την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων. Όμως αυτή η πρόταση της Κομισιόν παρουσιάζει διάφορα προβλήματα. Πρώτον, η επεξεργασία των υδάτων θα περάσει σε ιδιωτικά χέρια. Το είπε και ο ίδιος ο Επίτροπος. Καινούριε επιχειρηματικέ ευκαιρίε, είπε. Αυτοί βέβαια προφανώ, θα έχουν πιο πολύ στο μυαλό τους το επιχειρηματικό του συμφέρον και λιγότερο την υγεία μας. Σε ένα θέμα τόσο ευαίσθητο, ε, τα ύδατα θα πρέπει να παραμένουν σε δημόσιο, στο δημόσιο, σε κρατικά χέρια. Δεύτερον, αναγνωρίζεται ότι δεν θα μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε όλα τα ύδατα για ίδρευση όλων των καλλιεργιών. Οπότε η ερώτηση είναι, τα ύδατα τα οποία δεν θα χρησιμοποιηθούν για μια συγκεκριμένη καλλιέργεια, θα χρησιμοποιηθούν για κάποιες άλλες. Πώς θα εγγυηθούμε ότι δεν θα μολύνουν το υπέδαφος. Τρίτον, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κρύβουμε τα λίματά μας στις αγροτικές περιοχές. Οτιδήποτε φτάνει στο έδαφος μπορεί να καταλήξει τελικά στο ποτήρι μας ή στο πιάτο μας. Οπότε θα πρέπει να εργαστούμε επί άλλων μοντέλων ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Για τους πράσινους, ένα λεπτό, ο κ. Σκλέκ. Σκλέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε Βέλα, συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Μποναφέ για την εξαιρετική, τους έκθε, για την εξαιρετική της έκθεση. Με τις κοινέ μας προσπάθειες πετύχαμε μια πολύ καλά εξισορροπημένη έκθεση. Η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων έχει επιπτώσει στο περιβάλλον μας. Με την κακή διαχείριση του συστήματος μπορούμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στη σωστή χρήση των υδάτινων πόρων και στην τροφοδότησή μα, στην παροχή του νερού. Η έκθεση αυτή εντοπίζει σωστά αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να δούμε πώ θα περιορίσουμε τι αρνητικέ επιπτώσει στο περιβάλλον μα, το ίδιο και τη γεωργική παραγωγή. η γεωργία μπορεί να ωφεληθεί τα μάλα από την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λιμάτων, ιδίω τη νήσου. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε τι διάφορε παράγοντε μόλιν ρήπανση στο έδαφο, καθώ και την παρουσία μικροπλαστικών ή των ενδοκρινικών διαταρακτών στα επαναχρησιμοποιούμενα αστικά λίματα, ώστε να μην υπάρξουν άλλα προβλήματα υγεία. Ευχαριστούμε για την ΕΔΔ, κυρία Κοντά. Ευχαριστώ. Η έκθεση τη κυρία Μποναφέ είναι μια έκθεση κέρια, διότι προσφέρει συγκεκριμένε λύσει στα σοβαρά προβλήματα τη ε, σπάνιδος του νερού και της ε, ε, λειψιδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προβλήματα αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, ιδίω σε σχέση με την υπερθέρμανση του πλανήτη και τι κλιματικέ αλλαγέ. Ε, φύγουν το μεγαλύτερο μέρο των περιοχών τη Νότια Ευρώπη που κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν κρίση παροχή νερού και πίεση ω προ τροφο... το σύστημα τροφοδοσία του. Οι γεωργοί έχουν πληρώσει το τίμημα αυτή τη κρίση Καθώ τα συστήματα άρδευση πιέζονται. Θα πρέπει λοιπόν να πολλαπλασιαστούν οι καλέ πρακτικέ επαναχρησιμοποίηση των αστικών λιμάτων μετά τη συλλογή του, ε, προ το σκοπό τη άρδευση κυρίω. Είμαστε πολύ αποφασισμένοι να ελέγχουμε προσεκτικά την ποιότητα των νερών αυτών και να φροντίσουμε να μην υπάρχουν μικροπλαστικά και άλλοι ρηπογόνοι παράγοντε. Ε, εκεί θα πρέπει να υπάρχει τριπλή απέτηση να προστατεύουμε την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να εγγυόμαστε την σωστή τροφοδότηση σε νερό για όλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μελά για το ΙΕΝΕΦ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η πρόταση αυτή κανονισμού για την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λιμάτων ε, και των επεξεργασμένων λιμάτων ε, για σκοπού γεωργική χρήση είναι ένα θέμα μείζωνο σημασία για τρει βασικού λόγου, κατά την άποψή μα. Ε, με συγχωρείτε κυρία εισηγήτρια, είναι ψευδής είδηση ότι η ξηρασία και η έλλειψη νερού ε, αφορά την πλειοψηφία των περιοχών της Ευρώπης. Είναι ψευδής αυτές οι πληροφορίες που δεν αφορούν το σύνολο της επικράτειας, κυρίως έχουν να κάνουν με την ανεπάρκεια των εγκαταστάσεων και του συστήματος υδροδότησης. Γι' αυτό λοιπόν το ότι προτείνει η έκθεση αυτή είναι και την πόρτα στην διαχείριση άλλων, ε, από άλλους ε, των υδάτινων πόρων μας και όχι πλέον των κρατικών φορέων ή των υδάτινων ε, δημόσιων. Μας θυμίζει ένα τεράστιο σχέδιο όπως τα μεγάλα έργα που έγιναν στο 19ο αιώνα για την υδροδότηση. Η έλλειψη νερού για τους γεωργούς και τους κοινοτρόφους, η τεχνητή άρδευση και η, γεωπονική χημεία που θα είναι η στόχη του μέλλοντο θα μας κοστίσουν πολύ ακριβά. Θα μπορούσαν επίσης να είναι αντικείμενο ε, πολλαπλών κερδοσκοπικών προσπαθειών ή πολιτικών χειραγωγήσεων. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να ε, αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο και από το πρίσμα τη παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστούμε κύριο Λίζα για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε δικαίω πολύ αυστηρούς κανόνες για το πόσιμο νερό. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε τους ίδιους αυστηρούς κανόνες για όλες τις χρήσει νερού. Οπότε λογικό είναι να έχουμε μια κατάταξη. Η λειψιδρία είναι ένα θέμα, όχι μόνο στην Νότια Ευρώπη. Στη δικιά μου την περιοχή βρέχει κατά κανόνα πολύ και υπάρχει και μια παροιμία. Αν δεν θέλεις ε, να καείς διακοπές, ε, έλα στην ε, Ζάουρλαντ, γιατί βρέχει αλλά είναι η ε, λεκάνη απορροής και από εκεί που ιδρεύεται ολόκληρη η κοιλάδα του Ρουρ, 8 εκατομμύρια άνθρωποι. Λοιπόν, είχαμε πραγματικά όμως τέτοια ξηρασία και οι ταμιευτήρες ήταν ε, άδειοι και εκεί που λέγαμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε ποτέ πρόβλημα λειψιδρίας και δεν είχαμε ποτέ κανόνες βεβαίως σχετικούς, ε, ξαφνικά βρεθήκαμε με ζήτημα. Είναι λοιπόν και θέμα κλιματικής αλλαγής και θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί με αυτό το αγαθό. Οπότε θα πρέπει να είμαστε κάπως ε, πιο προσεκτικοί. Το ΕΛΚ θα ήθελε μια οδηγία και όχι κανονισμό για να είμαστε κάπως πιο ευέλικτοι στις επιθυμίες των ε, κρατών μελών, αλλά επί της αρχής είναι θετικό ε, το νερό το οποίο χρησιμοποιείται για ίδρευση να έχει βεβαίως αυστηρούς κανόνες αλλά όχι τους ίδιους με το πόσιμο νερό Ευχαριστώ λοιπόν όσου εργάστηκαν επί του θέματος και το ΕΛΚ θα στηρίξει το κείμενο αυτό. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό, κυρία Σάρμπου. Το έλλειμμα υδατοσυλληψιδρία ε, αποτελεί πρόβλημα για το 11% του πληθυσμού και το 17% της επικράτησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νερό είναι απαραίτητο για την παραγωγή τροφίμων, κατανοητικών αγαθών και ενέργειας. Για να προστατευτεί αυτός ο φυσικός πόρος είναι σημαντικό να βρούμε τις πιο κατάλληλες λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η οδηγία πλαίσιο για το ΙΔΟΡ αναφέρει την επαναχρησιμοποίηση ε, των αστικών λιμάτων ως έναν από τους ε, αποτελεσματικούς τρόπους ε, βελτίωσης αποδοτικότητας της διαχείρισης των υδάτων. Όμω ε, δεν έχουμε επαρκή νομοθετική στήριξη αυτής ε, της πρότασης. Η πρόταση της Κομισιόν δυστυχώ περιορίζεται στην χρήση αυτών των υδάτων στον γεωργικό κλάδο. Θα πρέπει οτιδήποτε γίνεται πάντως να γίνεται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η εισηγήτρια ζητά ένα κανονισμό για την εναρμόνιση της επαναχρησιμοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Κυρία Εύη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υποστεί πίεση και έλλειψη νερού λόγω των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και των κλιματικών αλλαγών. Η λειψιδρία έχει δημιουργήσει απώλειες τουλάχιστον 8,2 δις ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ιταλία ο αριθμός των ανθρώπων που πλήττονται από την ε, λειψιδρία είναι τουλάχιστον 20% με συνολικό κόστος το αστρομικό ποσό των 100 δις ευρώ. Όπω είπαν οι συνάδελφοι, αυτό αφορά την περίοδο ε, ξηρασία και ιδίω την λεκάνη τη Μεσογείου. Η λήψη δρία εντείνεται από τι κλιματικέ αλλαγέ και τι επιπτώσει του και πλήττει κυρίω το νότο τη Ευρώπη. Είναι αναμφίβολο λοιπόν το νερό ω κοινό αγαθό, ε, οικουμενικό αγαθό, είναι ένα πολύτιμο αγαθό και πρέπει να το ε, διαχειριζόμαστε με. Ε, σοφροσύνη θα πρέπει λοιπόν να βρούμε κοινού κανόνε για την επαναχρησιμοποίηση των αστικών λιμάτων στα πλαίσια τη κοινωνική οικονομία. Δεν μπορούμε παρά να τι δούμε θετικά. Ε, ο κανονισμό για την επαναχρησιμοποίηση είναι μια καλή ευρω... ευκαιρία που δεν θα πρέπει να τη χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξαμε τον ορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων για την συλλογή των ε, αστικών λιμάτων, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει ασφαλή επαναχρησιμοποίησή του. Δεν πρέπει να υπάρχει ποτέ κανένα κίνδυνο για το έδαφο και για τι καλλιέργειε. Κανένα περιθώριο για μικροπλαστικά και ενδοκρινικού διαταράκτε. Εδώ ήταν αποφασιστική η τοποθέτησή μα. Θα πρέπει αυτά να μην υπάρχουν καθόλου και στα νερά των ποταμών και των θαλασσών και κυρίω για να σεβόμαστε και τι προδιαγραφέ τη βιοπικιλότητα που διεθνώ ισχύουν. Θα πρέπει τα νερά που επαναχρησιμοποιούνται βάσει αυτού του κανονισμού να μπορούν όντω να επαναχρησιμοποιηθούν, ε, επιτρέποντα να σεβόμαστε και τι απαιτήσει υγεία. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και τι τοξικέ ε, ουσίε, όπω ε, φόσφορο, κάλιο και ούτω καθεξής. Αυτά δεν πρέπει να βρίσκονται ποτέ σε επαναχρησιμοποιημένα ύδατα. Γι' αυτό λοιπόν, αν είδη συμπεράσματο, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους κοιόδη εισηγητές για αυτόν τον τόσο σημαντικό κανονισμό. Και δύο λόγια για την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απειλεί την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε, κ. Λαντσίνη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να φροντίσουμε την προστασία των πολι... τη υγεία των πολιτών και του περιβάλλοντος. Θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας έναν κόσμο καθαρότερο και καλύτερο στι ε, μελλοντικέ γενιέ. Όμω χρειάζονται σταθμισμένε λύσει και μακροπρόθεσμε, χωρί απλώ να ξεκινάμε ένα κυνήγι μαγισσών με ξυπνάδε και ε, εφιολογήματα και να κοιτάξουμε ποια είναι η ορθή ε, προστασία του περιβάλλοντό μα. Ξέρουμε ποιε είναι οι πιέσει στην υδροδότηση που γνωρίζουν πολλέ περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε μια λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα και αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα πρώτο βήμα. Η επαναχρησιμοποίηση των αστικών λιμάτων είναι κάτι που θα μα επιτρέψει τουλάχιστον 6,7 κυβικά μέτρα, ε, δις μέτρα ε, εξοικονόμηση το χρόνο. Στην Ιταλία έχουμε ήδη κάνει κάποιε προσπάθειε και είδαμε ότι δεν υπάρχει μεγάλο κόστο για του γεωργού ω προ την άντρευση. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε προληπτικά ώστε η επαναχρησιμοποίηση των νερών να βασιστεί σε νέου κανόνε για όλε τι χώρε και αναρμονισμένα κριτήρια σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι προστατεύονται οι πολίτε και ότι υπάρχει καλύτερη ε, διάδοση των ορθών πρακτικών επαναχρησιμοποίηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Ντελαέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, κυρίε και κύριοι. Στο πλαίσιο τη λογική και κυκλική οικονομία, αυτή η έκθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μποναφέ και του συναδέλφου για τη δουλειά που έχουν κάνει. Πέραν το θέμα της διαφάνειας ευθύνη, ε, η ανάγκη της πρόθεσης της έρευνας και της καινοτοπία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ε, η υγειονομική κατάσταση των, των ε, κτημάτων μας, ε, των καλλιεργιών μας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί από την ποιότητα του νερού. Θα πρέπει οι γεωργοί να ενημερωθούν έτσι ώστε να χρησιμοποιούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα ανακυκλωμένα ύδατα και να μην επηρεαστούν από γενομικής πλευράς οι καλλιέργειές τους. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με τους καταναλωτές, οι οποίοι επίσης θα πρέπει να ενημερωθούν για να δεχτούν τη χρήση αυτού του ύδατος. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η πληροφόρηση και η επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων. Ευχαριστώ πολύ που η συγγήτρια δέχτηκε αυτές τις προτάσεις που έχω κάνει. Περνάμε στην διαδικασία Catch the Eye. Ποιος φαγιά. Πιο όμως αργά από την πρώτη φορά, ελπίζω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Από το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι η ξηρασία και η λειψιδρία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συστηματικά και συστημικά. Ε, πιο πρόσφατα, μέσω του προγραμματός δράσης για την κυκλική οικονομία, ξανασυζητήσαμε το θέμα αυτό. Τώρα η Κομισιόν ετοιμάζει το πρόγραμμα 2.0. Η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων κατόπιν εξερασίας τους για ίδρυυση θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ευτροφισμό στα ύδατα, είτε αυτά είναι στην επιφάνεια, είτε είναι υπόγεια. Και δεν θα πρέπει να πλήξει τη βιοπικιλότητα. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το ρόλο των αρμόδιων αρχών για, την, ε, για να βοηθήσουν το κοινό να συνειδητοποιήσει την ανάγκη χρήση επαναχρησιμοποίησης των υδάτων. είναι πολύ σημαντικό να γίνουν οι κατάλληλε επενδύσει. Ευχαριστώ πολύ. Κέλλη. Ε, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, το νερό πέφτει από τη βροχή, κυλάει στη θάλασσα, εξατμίζεται και ξαναγίνεται σύννεφο. Αλλά δεν είναι άπειρο. Έχουμε δει και περίοδους ε, ξηρασίας, ακόμα και στη χώρα μου που είναι γνωστή ως χώρα με πολλές ε, προκοπτώσεις. Ε, πέρσι το καλοκαίρι είχαμε όριο στη χρήση. Στο δε Δουβλίνο το μισό νερό χάνεται στους σωλήνες σύντρευσης και αυτό βέβαια πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η επαναξιμοποίηση των υδάτων όπου γίνεται είναι πάρα πολύ σημαντική και καλωσορίζω τις προτάσεις αυτές η Σιμώνα, η Μαριάννα, η Αντζελίκ, όλες αναφέρθηκαν στην ε, κυκλική οικονομία. Και βεβαίω εκεί πέρα εντάσσεται και η επαναξιμοποίηση του νερού. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μπορούμε να το επαναξιμοποιούμε και για ίδρυψη, άρδευση, οργία, Γιατί είναι ζωτική σημασία και πρέπει να το φροντίζουμε. Μια καλή πρόταση την οποία ευχαριστώ θα στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ολοκλώσαμε τη διαδικασία Κατστιάη. Κύριε κυρία Βέλα, έχετε το λόγο. Thank you, Madam President, and once again... Uh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω και την κυρία Μποναφέ για την επιτυχία της στην σύνταξη αυτής της έκθεσης και καλωσορίζω και τις ιδέες που υπέβαλαν ε, εδώ οι βουλευτές η Κομισιόν παρακολούθησε στενά την συζήτηση και θα εξετάσει λεπτομερώς τις προτάσεις του Κοινοβουλίου για να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα στην νομοθετική διαδικασία. Θα ήθελα όμως να αναφέρω κάποια πράγματα. Όσον αφορά τα μολυσμένα εδάφη, έχουμε την οδηγία περί αζωτούχων ακριβώς για να τα προστατεύσουμε και η Κομισιόν παρακολουθεί πολύ στενά την εφαρμογή αυτών των οδηγιών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να δικαιολογήσω το πώς ε, οι κακές ε, γεωργικές πρακτικές βλάπτουν τους ίδιους πόρους από ε, τους οποίους εξαρτάται η γεωργία. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι καμιά φορά υποτιμούμε το πρόβλημα όταν λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει λειψιδρία ο πλανήτης ολόκληρος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα και έτσι η αναγκαιότητα να δράσουμε άμεσα είναι ακόμη πιο επίγουσα. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, αν περιορίζεται σε γεωργία και άρδευση, θα ήθελα να πω ότι από τους διάφορους τομείς η γεωργία και η άρδευση είναι ακριβώς αυτή η οποία κάνει τη μεγαλύτερη χρήση νερού παγκοσμίω, όπως έδειξε και η μελέτη αντικτύπου έχει ακριβώς ε, τις περισσότερες δυνατότητες και υποχρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ λοιπόν η Κομισιόν συμφωνεί με την χρήση ανακυκλωμένου νερού, οι κανόνες αυτοί δεν αποκλείουν την δυνατότητα τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ε, το νερό αυτό και για άλλους σκοπούς. Είμαστε πεπισμένοι πως θα βρεθεί μια συμφωνία για τους νέους κανόνες και ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα την νομοθετική διαδικασία του πολύ σημαντικού αυτού φακέλου. Και το νέο αυτό μέσο θα διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό που υπάρχει με αυτήν την, τις δυνατότητες που μας δίνει αυτή η πρακτική και να χρησιμοποιήσουμε και τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα με ωφέλη και για τους γεωργούς, τους καταναλωτές και την ε, βιομηχανία. Η Κομισιόν λοιπόν αναμένει τις ε, διαπραγματεύσεις και είναι έτοιμη να στηρίξει τους ε, συνομοθέτες στην διαδικασία αυτή. Βασίζουμε όπως πάντα στην στήριξή σας και σας ευχαριστώ και πάλι για την προσήλωση που δείχνετε στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Τι συμβαίνει κυρία, κυρία μου. Κυρία Πρόεδρε, να θυμίσω στον κύριο Βέλε. Μπορεί να μας πει σήμερα κάτι παραπάνω για το πότε η οδηγία για τη μόλυνση στα δάφη θα είναι έτοιμη. Χθες δεν μου απάντησε. Ήταν βέβαια άλλο το θέμα, αλλά σήμερα θα ήθελα να έχω μια απάντηση. Κοιτάξτε, θα σα δώσω το λόγο σε ένα λεπτό. Απλώ να πω ότι κυρία Γκραπίνη δεν σα είδε κανεί. Δυστυχώ, παρόλο που ξέρουμε ότι συχνά συμμετέχετε στο Catch the τελείωσε η διαδικασία, δεν είχε γραφεί η παρέμβασή σα. Κύριε Βέλα, μπορείτε να απαντήσετε στην κυρία Γελαζέντερ και μετά να ολοκληρώσουμε την κυρία Μποναφέ. Κύριε Βέλλα, θα απαντήσετε στην ερώτηση της κυρίας Αγιάλα Σέντερ για το χρονοδιάγραμμα. Βέλλα, νομίζω έχει δίκιο η κυρία Βουλευτής. Πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια πρόταση για το πώς θα προχωρήσουμε. Την έχουμε συζητήσει την πιθανότητα, αλλά ως τώρα δεν έχει οδηγηθεί σε αίσιο πέρας η όλη κουβέντα. Ε, ελπίζω ότι θα γίνει σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Ελπίζω να δείξετε κατανόηση. Σας ευχαριστούμε κυρία Μποναφέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς οφείλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τα λόγια ε, ε, αυτά που εξέφρασε σήμερα, που δείχνουν την προσοχή του για το όλο θέμα, το ενδιαφέρον του, αλλά το έδειξε και από την αρχή τη θητεία του και μέχρι το τέλος του, ελπίζουμε. Το τέλος της θητείας του. Ευχαριστώ και του συναδέλφου που πήραν το λόγο, όχι μόνο για τη δουλειά των τελευταίων μηνών, αλλά και τα λόγια του σήμερα δείχνουν ότι στηρίζουν. Στηρίζουν την πρόταση αυτή, να πω σχεδόν ομόφωνα, ή τουλάχιστον Εβραίος. Σε κανέναν δεν διαφεύγει ότι το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό, θα έλεγα άκρο πολύτιμο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να σπαταλάμε ούτε ένα κυβικό μέτρο. Γι' αυτό λοιπόν και βάσει των αρχών τη κυκλική οικονομία, στην οποία βασίσαμε ολόκληρο το μοντέλο αναπτυξή μα στην Ευρώπη, θα πρέπει να ε, συμπεριλάβουμε και του υδάτινου πόρου. Οι αρχέ τη κυκλική οικονομία πρωτίστω επιβάλλουν την εξοικονόμηση ε, στη χρήση του νερού και την επαναχρησιμοποίηση. Επαναχρησιμοποίηση στη γεωργία και την κτηνοτροφία για σκοπού ε, αστικού, τον καθαρισμό των δρόμων, αλλά και βιομηχανικού. Βεβαίω, οπωσδήποτε έχοντα υπόψη τον πλήρη σεβασμό των κριτηρίων για την προστασία τη ανθρώπινη υγεία. Ε, αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα των κλιματικών αλλαγών. Εάν αυτή τη στιγμή δεν αλλάξουμε την πορεία μα ε, γοργά και με αποφασιστικότητα, θα πληγεί ανεπανόρθωτα το οικονομικό μα μοντέλο. Α προχωρήσουμε λοιπόν με τη σωστή χρήση των υδατινών πόρων, με τα μέτρα αυτά που θέλουμε να εγκρίνουμε στο δυνατόν νωρίτερα και με τι απαραίτητε επενδύσει στον τομέα αυτό. Διότι για την ορθή διαχείριση των υδατινών πόρων χρειάζονται βεβαίω και ε, σοβαρέ επενδύσει. Ευχαριστούμε πολύ. Η συζήτηση λοιπόν κλείνει. Η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα αργότερα σε περίπου 13 λεπτά μικρή διακοπή της Συνόδου μέχρι τότε.

Uh, Συναδελφοι, Αδελφοί, παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις ψηφοφορίες. Παρακαλώ καθίστε, ξεκινάμε. So, colleagues, uh, the first we vote on... Λοιπόν, συνάδελφοι, ψηφίζουμε πρώτα απ' όλα στην Συμφωνία Σύμπραξη Σύμπραξης ε, με την ακτή του Ελεφαντοστού, έκθεση Φεραίρα, άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερη ψηφοφορία, το ψήφισμα της έκθεσης Φερέρα. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην συμφωνία με το Μαρόκο. Έχουμε το αίτημα του συναδέλφου Μαρσελιέζη, ο οποίος θέλει να μιλήσει σύντομα. 30 δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η Human Rights Watch μας ενημερώνει, μας προειδοποιεί ότι ψηφίζουμε ε, μία συμφωνία αλίας με το Μαρόκο που ε, προσβάλλει τα διεθνή, το διεθνές δίκαιο. Ε, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε υπεράνω των νόμων. Θα έπρεπε να ζητήσουμε καταρχήν τη γνωμοδότηση του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο, μας ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ γιατί να μην μα ενδιαφέρει και αλλού στον κόσμο. Θα έπρεπε να ζητήσουμε πρώτα τη γνωμοδότηση τη Δικαστήριου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Thank you. And now we can proceed to the vote. Ευχαριστώ. Περνάμε στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το ψήφισμα σύνολο του υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θα το επαληθεύσουμε βεβαίως. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην έκθεση Καντέκ ε, για την ε, συμφωνία με το Μαρόκο. Με ονομαστική ψηφοφορία σας παρακαλώ, πρόκειται για σύμφωνη γνώμη. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρασε Και εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση Νικολάη για την αποτροπή της αναρχής αλληλείας στον κεντρικό Αρκτικό ωκεανό. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Μετά έχουμε την έκθεση Ροντρίγκε Πινέρο το πρωτόκολλο στην Συμφωνία για την Οικονομική Εταιρική Σχέση της Ευρωπαϊκής Σχέσης και του Μεξικού για την προσχώρηση της Κροατίας. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μετά. Έκθεση Σαλαφράνκα Έχουμε τις ε, τροπολογίες της Επιτροπής Αμπλοκ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά. Τροπολογία 45D με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δι με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται μετά 37 έως 38 της Επιτροπής υπέρ κατά άποχες εγκρίνονται μετά ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση της Κομισιόν άρχεται η ψηφοφορία και πέρας και εγκρίνεται τώρα Ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περνάμε σε μια άλλη έκθεση του συναδέλφου Καντέκ. Το πολιετέ σχέδιο για τα αποθέματα υγδίων στα δυτικά ύδατα, παρακείμενα ύδατα και αλληλευτικέ δραστηριότητε εκμετάλλευση. Έχουμε την 99 τη προφορική συμφωνία. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μετά. Κοινή δήλωση τροπολογία 100 της Επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωση. Μετά. Έκθεση Γκαρντίνη. Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης. Τροπολογία 79 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Μετά έχουμε την κοινή δήλωση τροπολογία 80 της Επιτροπής υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και άρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ε, πρώτης ανάγνωσης. Περνάμε στην έκθεση Μποναφέ ελάχιστες απαιτήσει για την επαναξιμοποίηση των υδάτων ψηφίζουμε πρώτα απ' όλα τις τροπολογίες αρμόδιας επιτροπής unblock υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 121 της επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές να το δούμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μετά. Τροπολογία 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μετά την 90 της Επιτροπής. Τι θέλετε, να την επαληθεύσουμε την 135. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 90 της Επιτροπής υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε την πρόταση της Κομισιόν με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται και άρα ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση περνάμε στην πρώτη έκθεση ε, της ε, κυρίας, ε, του κυρίου Ντάντη. Έγκριση και υποπτήρια της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων. Ψηφίζουμε το τροπολογία 4 προσωρινή συμφωνία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και πάλι ολοκληρώθηκε εδώ η πρώτη ανάγνωση. Δεύτερη έκθεση του κυρίου Ντάντη πρόγραμμα για ενιαία αγορά ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων ε, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω τον λόγο στον εισηγητή. Έχει τον λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά συγκεντρώνει 7 υπάρχοντα προγράμματα και προβλέπει νέα μέτρα ε, εναρμονισμένα για την ενίσχυση τη ενιαία αγορά. Μιλάμε για ε, χρηματοδότηση που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περίοδο 2021-2027, ώστε να υποστηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα του μηχανικού μα κλάδου, ιδίω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ε, ε, μικρών, την στήριξη της διατροφικής αλυσίδα, την υγεία των ανθρώπων, ζώων και φυτών, την καλύτερη προστασία των καταναλωτών, καθώς και τη δημιουργία πλαισίου για την χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών στατιστικών ε, μελετών. Ε, ο στόχος που πετύχαμε είναι πολύ φιλόδοξος και προβλέπει αυτή τη στιγμή ως προς μια, μια συνολική μάλλον πρικοδότηση 6 δι, εκ των οποίων τα 3 δι προβλέπονται για το κόσμο, για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, που είναι ο βασικότερο άξονα του οικονομικού συστήματο ε, και τη παραγωγή στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα κονδύλια προβλέπονται για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων παρακολούθηση τη ε, αγορά και τη ασφάλεια των προϊόντων, με ιδιαίτερη προσοχή στα προϊόντα τα οποία πολλούνται online. Επιπλέον, η κατεξουσιοδότηση ε, πράξεων για την υλοποίηση του προγράμματο επιτρέπουν την άσκηση ελέγχου από το Κοινοβούλιο. Με το κείμενο που θα εγκρίνουμε, συνάδελφοι, το Κοινοβούλιο τοποθετείται ξεκάθαρα και με φιλοδοξία υπέρ του παραγωγικού συστήματος στην Ευρώπη και υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχόμεθα και το Συμβούλιο να δείξει την ίδια διάθεση. Ευχαριστούμε. Thank Σας ευχαριστώ. Ψηφίζουμε τώρα την πρόταση για να απορριφθεί η πρόταση της Κομισιόν. Τροπολογία 150 υπέρ. Κατά. Αποχές πρόταση απόρριψης πρότασης Κομισιόν απορρίπτεται. Μετά περνάμε στο σχέδιο του νομοθετικού κειμένου. Έχουμε τις ε, τροπολογίες των μελών τη Επιτροπή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία από την Αρμόδια Επιτροπή χωριστές. 25 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές να την απαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται ναι, την πλειοψηφία δεν το είχα δει συγγνώμη 38 της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 της Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά με ονομαστική ψηφοφορία 154 άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 δι με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα. Ε, τροπολογία 1 της Επιτροπής ΠΕΡ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά. 152 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. απορρίπτεται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα η πρόταση της Κομισιόν με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται και τώρα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση ψηφίζουμε τώρα την έκθεση του συναδέλφου Μαρτουσέλο. Ψηφίζουμε τις ε, τροπολογίες επί τα επιτροπής υπέρ κατά εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 29 της Επιτροπής υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την πρόταση της Επιτροπής. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Και πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο ψήφισμα για την ένταξη των Ψηφίσαμε το αρχικό κείμενο 2. Ψηφίζουμε τη 2.4 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 2, σημείο 6. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3, σημείο 4 το αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3 μετά το σημείο 4. Θα δώσω το λόγο στην κυρία για μια προφορική τροπολογία. Παρακαλώ. Ως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για ε, το θέμα των δικαιωμάτων των Ρωμά ε, θεωρώ ότι θα πρέπει τα παιδιά να είναι προτεραιότητα στην εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για τους Ρωμά. Είναι σημαντικό να προστατέψουμε και να προωθήσουμε την ίση πρόσβαση σε όλα τα δικαιώματα από, τα, από πλευράς όλων των παιδιών Ρωμά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κορατσαμπίλ. Υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι. Την ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, Β της αιτιολογικής έκθεσης, αρχικό κείμενο, σε εξηγωστή ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα ας ψηφίσουμε το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προχωράμε. Εκθέση τη κυρία Μπαγκατσαουρουτούντου Αρούη. Εφαρμογή των διατάξεων τη συνθήκη που αφορούν την ηθαγένεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίζουμε τροπολογία 4. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. The vote is Απορρίπτεται. 6. Το αρχικό κείμενο. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Λίγη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Λίγη. Απορρίπτεται. Περνάμε στο αρχικό κείμενο τώρα, ονομαστική ψηφορία ε, για την παραφωνιά. Άρχεται, λίγη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7, ονομαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Και πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Λίγη. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο της παράγραφου 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 30 σε δύο τμήματα το αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επαληθεύουμε την παράγραφο 30 δεύτερο τμήμα. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 38. Το αρχικό κείμενο. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Παράγραφος 39. Από το αρχικό κείμενο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 42 το αρχικό κείμενο, Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Υπέρ, υπέρ λέω. Κατά. εποχές... Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. εποχές... Εγκρίνεται. Παράφος 46. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. εποχές... Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Δεύτερο τμήμα της παράγραφου 46. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει. Λίγη. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Με ονομαστική ψηφοφορία και πάλι. Άρχεται. Λίγη. Απορρίπτεται. Παράγραφος 49 του αρχικού κειμένου με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 και πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη. Απορρίπτεται. Παράγραφος D της αιτιολογικής έκθεσης τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στο αρχικό κείμενο του D σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ας ψηφίσουμε στο σύνολο του κειμένου του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη. Λήξη.